Uh, Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Προτείνω να ξεκινήσουμε, διότι έχουμε εδώ την Επίτροπο Καντή Σίμψον, που είναι Επίτροπος για την Ενέργεια, για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που μας περιμένει. Θέλω λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε κάθε ευκαιρία και όλο το χρόνο για να έχουμε καρποφόρο ο διάλογο σιγά σιγά όσο περνάει η ώρα σίγουρα θα έρθουν και άλλοι συνάδελφοι στην αίθουσα. Λοιπόν, καλωσορίζω την κυρία Κάντρι Σίμψον, η οποία δέχτηκε την πρόσκλησή μας να έρθει εδώ στην Επιτροπή μας για ανταλλαγή απόψεων, κυρίως για τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος. Θέλω να επενθυμίσω στα μέλη ότι η κατεξοδότηση ε, πράξη ε, έφτασε στο Κοινοβούλιο την 31η Οκτωβρίου για έλεγχο. Και η Επιτροπή μας αποφάσισε να επεκτείνει την περίοδο για δύο επιπλέον μήνες και να ξανακαλέσει την Επίτροπο εδώ για παρετέρω συζητήσεις. Έχουμε στη διάθεσή μας λοιπόν μια μισή ώρα για τη συζήτηση αυτή, μέχρι τις 10 και 30. Και με τη βοήθεια των διερμηνέων θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και εύχομαι να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα αυτό το χρόνο. Θα ζητήσω λοιπόν από την κυρία Επίτροπο πρώτα απ' όλα να μας παρουσιάσει μια σύντομη εισαγωγή, 10 λεπτά, και μετά θα ακούσουμε τους συντονιστές ή τους αναπληρωτές τους για ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων. Στη συνέχεια θα ακούσουμε απαντήσεις από την Επίτροπο και μετά υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν καταγραφεί στον κατάλογο ομιλητών για να πάρουν το λόγο στη συνέχεια και θα έχουμε και δεύτερο γύρο. Ένα λεπτό καθένας όμως θα είναι στον τελικό γύρο και θα έχετε φυσικά και εσείς τη δυνατότητα να απαντήσετε και να έχουμε και έναν επίλογο. Λοιπόν, ζητώ από την Επίτροπο να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, καλημέρα. Ευχαρίστως να ξεκινήσω. Είναι η πρώτη μου φορά ως ε, νέα επίτροπος. Και πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ και εσάς. Ε, νομίζω ότι και για τους δυο μας είναι ένα νέο ξεκίνημα αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκλησή σας. Για αυτή την ανταλλαγή απόψεων για τον ενωσιακό αυτοκατάλογο κοινών έργων. Όπως έλεγα, είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψε, απόψεων που έχουμε μεταξύ μας από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, αυτή τη βδομάδα μόλις, και θέλω έτσι να αποτελέσει μια κίνηση για να συνεχή διάλογο μεταξύ μας όσον αφορά θέματα ενεργειακής πολιτικής και νομίζω ότι σας το έχω ήδη δείξει ότι είμαι ανοιχτή για συνεργασία μεταξύ μας. Νοέμβριος 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την ε, προβολή της για μια οικονομία η οποία να είναι σύγχρονη, να βοηθάει στην ευημερία, να είναι ανταγωνιστική και ουδέτερη όσον αφορά το κλίμα, με φιλόδοξους ε, στόχους για το 2050. Είδε την επόμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την ηγεσία βέβαια της Προέδρου Ούρσουλα von der σκοπεύει να ανακοινώσει τις δεσμεύσεις αυτές πιο συγκεκριμένα και να ξεκινήσει με το περίφημο European Green Deal, την πράσινη συμφωνία δηλαδή, που αποτελεί και μια εμβληματική πολιτική πρωτοβουλία. Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι μας, και εσείς δηλαδή, θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για αυτήν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι Μόνο τα πλαίσια μπορώ να βάλω για την συζήτηση, γιατί είναι η ίδια η πρόεδρος Φόντερ Λάιεν, η οποία θα παρουσιάσει την πρωτοβουλία αυτή την επόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή που έχουμε την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια να σας παρουσιάσει την Πράσινη Συμφωνία, η οποία ε, αλλάζει την Ευρώπη, την κάνει περισσότερο καθαρή, που να χρησιμοποιεί τους σπόρους πιο αποτελεσματικά ε, με μια κοινωνία και οικονομία περισσότερο ανταγωνιστικές. Είναι μια πολύ καλή στρατηγική που θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, ε, νέες θέσεις απασχόληση, θα χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες και θα φροντίσει η πυρός μας να είναι κλιματικά ουδέτερη το 2050 το μερίδιο του ηλεκτρισμού θα διπλασιαστεί σε σχέση με τώρα όσον αφορά ε, τους πόρους που θα χρησιμοποιούμε για αυτόν, που θα είναι κυρίως ηλιακή και η ολική ενέργεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν και υποδομές κατάλληλες, σύγχρονες, ασφαλείς και ε, που να λειτουργούν με φύ ενέργεια για αυτήν την ενεργειακή μετάβαση. Να είσαστε σίγουροι λοιπόν ότι η ασφάλεια εφοδιασμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά αποτελούν προτεραιότητα για μας. Τώρα, τα προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος έχουν αποδειχθεί πάρα πολύ σημαντικά για τα διασυνδεόμενα ενεργειακά δίκτυα. Από το 2014 η πολιτική μας για τα ενεργειακά δίκτυα έχει δώσει αυτά αποτελέσματα με συγκεκριμένα προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος, ώστε να μην βρίσκονται στην απομόνωση κάποιες ευρωπαϊκές περιοχές, από τη Μάλτα μέχρι την Φιλανδία, και προκειμένου να υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός στις αγορές μας και να χρησιμοποιούν περισσότερο νόσιμες πηγές. Η πολιτική μας επίσης επέτρεψε στην Ευρώπη να προχωρήσει σε 30 ε, βασικές ενεργειακές υποδομές και με 75 επιπλέον ε, προγράμματα που αναμένονται να υλοποιηθούν μέχρι το 2022. Όλα αυτά βοηθούν τις χώρες μέλη να πετύχουν το 10% ε, διασύνδεση με ηλεκτρικά δίκαια, δίκτυα μέχρι το 2020 και 15% μέχρι το 2030. Ο κύριος Κανιέτε τον ε, Οκτώβριο μας είχε αναφέρει τα διάφορα προγράμματα. Ο νέος κατάλογος αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στα συστήματα ηλεκτρισμού. Χρησιμοποιείται όλο περισσότερο ο ηλεκτρισμός και επίσης χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ενώσιμες πηγές ενέργειας για την παραγωγή του. Αυτές ε, οι νέες επενδύσεις όμως θα πρέπει να πάνε χέρι-χέρι με την ψηφιοποίηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δράσει από πριν προκειμένου να μειώσει τον αριθμό των προγραμμάτων που βασίζονται στο φυσικό αέριο. Και ο πρώτος κατάλογος, από ό,τι ξέρω, είχε 107 τέτοια προγράμματα φυσικού αερίου. Ε, το τρίτο, ο τρίτος κατάλογος θα έχει 53. Και έχουμε ήδη προχωρήσει πάρα πολύ με 32 τέτοια προγράμματα φυσικού αερίου που περιλαμβάνονται στον τέταρτο κατάλογο. Και τώρα προχωρούμε ακόμα περισσότερο υπέρ της ενεργειακής ε, ασφάλειας και προκειμένου να υπάρχει διαφοροποιημένος εφοδιασμός. Όταν ε, λοιπόν ε, μέχρι το 2020 θα έχουν υλοποιηθεί τα ήδη τρέχοντα προγράμματα, όλες οι χώρες θα έχουν πρόσβαση σε τρεις τουλάχιστον πηγές φυσικού αερίου ή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Είναι επίσης σαφές ότι προσλέπουμε στον στόχο του 2050 για ε, ουδετερότητα όσον αφορά το κλίμα. Οπότε, οτιδήποτε παραμένει στην Ευρώπη από φυσικό αέριο θα πρέπει να εξαφανιστεί σιγά σιγά. Ε, αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι υπάρχουν και ανησυχίες. Αλλά να ξέρετε ότι δουλεύω χωρίς σταματημό για να αντιμετωπίσω ό,τι δυσκολίες προκύπτουν. Έπειτα, η αναθεώρηση των ε, διευρωπαϊκών ε, δικτύων και ο σχετικό κανονισμό είναι προτεραιότητά μου για το 2020. Έχω ζητήσει αξιολόγηση και περιμένω προτάσει και από του συνομοθέτε μέχρι τα τέλη τη επόμενη χρονιά το έργο μας πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα για να πετύχουμε τους ε, στόχους μας, τους ενεργειακούς και τους κλιματικούς, έτσι όπως συμφωνήθηκαν στο Παρίσι, προκειμένου να έχουμε ε, μια Ευρώπη καθαρή όσον αφορά την ενέργεια. Στόχος μου είναι λοιπόν να συνεχίσω να στηρίζω την ενεργειακή μετάβαση και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Επίσης εργάζομαι σκληρά για να έχουμε ένα νέο πλαίσιο για τα διευρωπαϊκά δίκτυα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν μπορώ βέβαια να σταματήσω μέχρι να τα καταφέρω. Μας ζητήθηκε να φτιάξουμε ένα κατάλογο PCI κάθε δύο χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε τον πέμπτο τέτοιο κατάλογο έτοιμο προς έγκριση για το 2021. Η διαδικασία για να προετοιμαστεί ο κατάλογος είναι μια διαδικασία που κρατάει δύο χρόνια και ήδη ξεκινήσει βασιζόμενοι στο σημερινό πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν με την κατάρτιση του πέμπτου καταλόγου με τους τρέχοντες κανόνες, αλλά σίγουρα μπορούμε ήδη να κάνουμε πολλά ώστε να εκφράσουμε στο νέο κατάλογο τις κλιματικές μας φιλοδοξίες. Τι μπορούμε να κάνουμε ήδη. Πρώτον, μπορούμε σημαντικά να βελτιώσουμε την αξιολόγηση βιωσιμότητα όλων των υποψηφίων προγραμμάτων φυσικού αερίου και έχω ζητήσει από τι υπηρεσίε μου να θέσουν σαφή κριτήρια μέχρι τα μέσα του 2020. Δεύτερον, θα προσπαθήσω να ενσωματώσω περισσότερα προγράμματα ενεργειακής μετάβασης στη διαδικασία αυτή εκπόνησης του καταλόγου. Αυτό σημαίνει ε, έξυπνα δίκτυα και προγράμματα υποδομών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και καινοτόμα προγράμματα. Όλα αυτά τα προγράμματα επιτρέπουν την ε, μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας και την απαλλαγή από τον άνθρακα. Τρίτον, είμαι έτοιμη να ενισχύσω περισσότερο τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να δημιουργήσω έναν συνεχή πολιτικό διάλογο που θα βασίζεται στις πρακτικές όπως καθόρισε ήδη ο προκάτοχός μου ο κύριος Αρίας Κανιέτε. Είμαι έτοιμη λοιπόν για συζητήσεις με την Επιτροπή σας Ήτρε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έχουμε τον εντοπισμό των υποδομών που χρειάζονται σε κάθε ευρωπαϊκή περιοχή, όπως επίσης και την αξιολόγηση των υποψηφίων προγραμμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν και έτσι να δώσουμε νέες ευκαιρίες σε όλους. Να ξέρετε ότι θα ζητήσω τη συμμετοχή της Επιτροπής Ήτρε και για την κατάρτιση του 5ου καταλόγου PCI. Με όλα αυτά κατά νου λοιπόν βασίζομαι στη στήριξή σας και για τον 4ο κατάλογο PCI. Είναι ο μόνος ο τρόπος να προχωρήσουμε γιατί πρέπει με νέο πνεύμα να προσαρμοστεί ο κατάλογος ώστε να έχουμε καλύτερα περισσότερο αντοχής και πιο ικανοποιητικά για όλους ενεργικά συστήματα. Πρέπει να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε αποτελέσματα, φιλόδοξα αποτελέσματα και ένα νέο πλαίσιο για τις αυριανές ενεργειακές υποδομές. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you very much, Commissioner. Επίτροπε, ευχαριστούμε που ήρθατε. Για την... Ευχαριστούμε για τη δέσμευσή σας. Να συνεισφέρετε κι εσείς μαζί με άλλους συμφεροτούχους στην... στο μετασχηματισμό των ενεργειακών συστημάτων για να πετύχουμε τους στρατηγικούς μας στόχους. Την επόμενη εβδομάδα είναι η εβδομάδα της Πράσινης Συμφωνίας. Η εβδομάδα που θα παρουσιάσετε την Πράσινη Συμφωνία. Ε, μιλάμε για την αναθεώρηση του τρέχοντος κανονισμού για να έχουμε ένα νέο πλαίσιο για έργα κοινού ενδιαφέροντος. Σημαντικό αυτό που είπατε, ότι στο μέλλον θα προσπαθήσετε να συμπεριλάβετε στον κατάλογο περισσότερα ενεργειακά προγράμματα μετασχηματισμού. Το Κοινοβούλιο θα σας στηρίξει όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά και για άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, θα δώσω το λόγο στους συντονιστές. Ο κύριος Λέναρτ από το ΕΛΚΑ είναι ο πρώτος. Καλώς ήρθατε, Επίτροπε, στο Κοινοβούλιο. Πρώτη φορά έρχεστε εδώ. Χαιρόμαστε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Να πω ευθύς εξ αρχής ότι πάντα πιστεύουμε ότι οι τρεις στόχοι της βιωσιμότητας, ενεργειακής ασφάλειας και ε, προσπελάσιμων τιμών είναι κέρυοι στόχοι. Αυτή είναι η πραγματική στόχη Ε, για τις μεταδοτικές φιλοδοξίες για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα ε, συμφωνούμε. Θεωρούμε ότι οι διασυνδέσεις των αγωγών φυσικού αερίου σε μια μεταβατική φάση ως κρίσιμη σημασία για να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους της μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα. Ιδίω και αυτή είναι μία από τις φιλοδοξίες που υπάρχουν και στα ερευνητικά προγράμματα και στα οποία συμφωνήσαμε με την ε, με τις υπηρεσίες σας και άλλες γενικές διευθύνσεις σε διαπραγμάτευση με το Κοινοβούλιο, εάν θέλετε να έχετε ε, έργα χωρίς α, διοξείδιο του άνθρακα. Χρειάζεστε αυτή την υποδομή του φυσικού αερίου για το μεθάνιο. Χρειάζεται, χρειάζεστε φυσικό αέριο στην αρχή για το μπλε υδρογόνο. Γιατί ναι, κανονικά θα πρέπει να είναι πράσινο υδρογόνο, αλλά αν θέλουμε τα επόμενα δύο χρόνια να έχουμε ε, χαλιβουργίες, ας πούμε, ε, χωρίς καθόλου διοξίδιο του άνθρακα, χρειαζόμαστε ε, το φυσικό αέριο ως βασική τεχνολογία, ως βάση ε, στη φάση που το μεθάνιο υποκαθιστά το χάλιβα. Τον άνθρακα, συγγνώμη, τον άνθρακα. Πρόσφατα συγκεντρωθήκαμε οι 41 περιοχές που παράγουν άνθρακα στην Ευρώπη και που βρίσκονται σε μετάβαση. Και οι εκλογές σε, αυτή την, σε αυτές τις περιοχές, όταν έγιναν εκλογές λοιπόν, ε, όλοι οι ψηφοφόροι πήγαν και ψήφισαν ακραία κόμματα. Τα δημοκρατικά κόμματα έχασαν 100%. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε ένα δημοκρατικό project. Όχι να μειώσουμε τις φιλοδοξίες ό,τι αφορά τη μείωση του του άνθρακα, αλλά μιλάμε για ένα περίπλοκο πλαίσιο, όχι μόνο να μειώσουμε δηλαδή το διοξείδιο του άνθρακα, το θέμα είναι πώς θα το κάνουμε αυτό. Ε, τα λεφτά από τον ορίζοντα 2020 ε, θα επενδυθούν για να μειώσουμε ακριβώς ε, το διοξίδιο του άνθρακα, αλλά για, να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχουμε σαν βάση το φυσικό αέριο. Πρέπει να έχουμε την κατάλληλη υποδομή, δηλαδή, φυσικού αερίου. Για μας, ως ΕΛΚ, είναι πολύ σημαντικό και συμφωνούμε με την μεταρρύθμιση των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας, αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε τους τρεις στόχους που είπα στην αρχή και να έχουμε και την τεχνολογία του φυσικού αερίου ως βάση. Αλλιώς δεν πρόκειται να το πετύχουμε αυτό, να πετύχουμε τη μείωση δηλαδή ε, του διοξιδίου του άνθρακα σε ενεργοβόρες ε, επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε την υποδομή του φυσικού αερίου για να τα καταφέρουμε. Αλλά καταλαβαίνετε, θέλουμε να μειώσουμε το διοξίδιο του άνθρακα ε, και θέλετε, ας πούμε, στε χαλιβουργίες να μειωθεί αυτό το διοξίδιο του άνθρακα και παράλληλα λέτε ότι πρέπει να μειώσουμε και το φυσικό αέριο. Δεν γίνονται αυτά μαζί. Ο κ. Γκονζάλες Θέσαρες. Ε, καλώς ήρθατε, Επίτροπε. Και καλή επιτυχία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία και ελπίζω να υπάρχει καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή μας. Για αυτό το έργο κοινού ενδιαφέροντος θα πρέπει να δούμε πώς καταρχάς λειτουργούμε σε αυτή την Επιτροπή. Ε, υπάρχει ο πέμπτος κατα... Δεσμευτήκαμε να φτιάξουμε τον πέμπτο κατάλογο σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Εσείς δεσμευτήκατε. Αυτός ο κατάλογος Ελπίζω να μην μας το φέρετε έτοιμο την προηγούμενη μέρα και μας πείτε αυτός είναι, χωρίς δυνατότητα συνεργασίας επί του καταλόγου. Είναι σημαντικό να δούμε ένα προσχέδιο. Το είχε, είχε δεσμευτεί ο κύριος Κανιέτε απέναντι στην Επιτροπή μας και στην ομάδα μας ότι θα δουλέψουμε μαζί για την εκπόνηση του καταλέγου. Ελπίζουμε να τιμηθεί αυτός, αυτή η δέσμευση και να μην μείνουν ας πούμε, λόγια και ένα περιεχομένο, αυτά που είχε πει ο Επίτροπος Κανιέτε. Όπως είχα πει και στην πρώτη παρουσίαση του τετάρτου καταλόγου των έργων κοινού ενδοεφέροντος, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο κατάλογος των ΕΚΕ. Για δύο λόγους. Καταρχάς, δείχνουν το πώς θα προχωρήσει η Ευρώπη της ενέργειας και πώς θα βελτιώσουμε την ασφάλεια ανεφοδιασμού. Και θα μας επιτρόψει να μειώσουμε την ε, τιμή της ενέργειας για όλους τους πολίτες και θα πρέπει να διευκολύνουμε την, ε, την οικολογική μετάβαση και τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό το τελευταίο σημείο μας απασχολεί, γιατί θα πρέπει, υποτίθεται, να, να χρηματοδοτήσουμε υποδομές ε, αμφισβητούμενες μέχρι το 2050 που θα μπορούσε να μπλοκάρει την ε, τεχνολογική εξέλιξη ενός συστήματος που είναι ουδέτερο σε διοξίδιο του άνθρακα. Ξέρουμε ότι το φυσικό αέριο, το χω, χωρίς διοξείδιο του άνθρακα θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο, αλλά δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε με τεχνολογίες μέχρι το 2050 που είναι ασύμβατες με την ουδετερότητα αυτή. Δεν έχουμε στοιχεία για να ε, μελετήσουμε την επίπτωση αυτών των έργων. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, Επίτροπε, μπορείτε να μας εξηγήσετε η ε, ισορροπία ανάμεσα σε έργα ε, ηλεκτρική ενέργειας και φυσικού αερίου, πώς εξασφαλίζεται στον κατάλογο. Και τα έργα φυσικού αερίου, ε, τι, πώς παντρεύονται με το φυσικό αέριο άνευ διοξιδίου του άνθρακα. Τι συμβατότητα έχει αυτός ο κατάλογος με, το, με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που θα μας παρουσιάσετε την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια πριν παρότι θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα. Επίσης, ε, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων για την χρηματοδότηση ε, προγραμμάτων και έργων που έχουν να κάνουν με τα ορικά καύσιμα. Τι επίπτωση θα έχει αυτή η απόφαση στην, ε, στον τέταρτο κατάλογο και στον πέμπτο κατάλογο, αν μπορείτε. Επίσης, ο Γενικός διευθυντή για την Ενέργεια είπε ότι πρέπει στο μέλλον να μεταρρυθμίσουμε σωστά τον κανονισμό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα για να τα προσαρμόσουμε ε, με, τα, με τους στόχους για την μείωση της κλιματικής αλλαγής. Κομισιόν, τι θα κάνετε την επόμενη χρονιά ε, σε αυτή την προσπάθεια μεταρρύθμισης. Όσο γρηγορότερα ξεκινήσουμε την προσπάθεια αυτή, τόσο καλύτερα. Γιατί δεν είναι εύκολη προσπάθεια. Ευχαριστούμε, Επίτροπε, και καλή τύχη. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Από το ο κύριος Πετέρσεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο. την Επίτροπο. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας σήμερα. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον κύριο Μπόχρα πριν από κάποιε εβδομάδε το συγκεκριμένο θέμα. Είναι λοιπόν εξαιρετικό το ότι έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και μαζί σα σήμερα. Στην προηγούμενη θητεία εργαστήκαμε σκληρά για να προσπαθήσουμε να ενοποιήσουμε την αγορά σε όλη την Ευρώπη. Αγορά ηλεκτρισμού, έχουμε οδηγίε, κανονισμού, ε, το κανονισμό Acer. Έχουμε πάρα πολύ καλά εργαλεία για να ενοποιήσουμε περαιτέρω τις αγορές. Γιατί δεν υπάρχει πραγματική ενιαία αγορά σε ό,τι αφορά την ενέργεια σήμερα. Άρα, θα πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε τους πόρους μας παντού. Και προφανώς τα PCR είναι πάρα πολύ σημαντικά σε ό,τι αφορά την περαιτέρω ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς. Ως εκ τούτου Προφανώς και παίζονται μεγάλα συμφέροντα εδώ. Θέλουμε να εναρμονίσουμε φυσικά αυτά που κάνουμε εδώ και τις αποφάσεις που λαμβάνουμε με τους στόχους του Παρισιού. Και γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο σημαντικός ο κανονισμός αυτός. Και με ενθάρρυναν αυτά που είπατε σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού, αλλά θα σας καλούσα να υποβάλλετε ένα πιο φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα, εφόσον είναι δυνατόν, δεδομένου και αυτά που είπατε για την παρουσίαση της Πράσινης συμφωνία. προκειμένου να μπορέσουμε να πάμε στην COP25 με μια σαφή φιλοδοξία να καθιστούμε φιλο, ουδέτερη όσο τον άνθρακα μέχρι το 2050 και αυτό θα πρέπει να συνάδει με όλου του στόχου σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Και προφανώς με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία ανέφερε ο συνάδελφος ο κ. Έιλερ, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην επενδύσουμε σε πόρους οι οποίοι στην τελική ανάλυση να καταστούν παροχημένοι. Άρα, σας απευθύνω έκλεξη να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό και να υποβάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα πιο φιλοδόξο. Και κατά δεύτερον, νομίζω ότι καλό θα ήταν να υπάρχουν αξιολογήσει ε, του αντικτύπου στο περιβάλλον σε ό,τι αφορά τις επενδύσει αυτές. Αυτός ε, θα μπορούσε να συνεπάγεται πιο ε, μεγάλο ρόλο και τον είστε στο σημείο αυτό. Και εδώ λοιπόν θεωρώ ότι έχει ρόλο να παίξει θα ήταν χρήσιμο αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του αντικτύπου στο περιβάλλον. Και τέλος, να δούμε τι γίνεται με τον εναρμονισμό των PCI σε ό,τι αφορά με αυτά που γίνονται στην ΕΤΕΠ. Όλα αυτά προχωράν γρήγορα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ενήμεροι στην αναθεώρηση του κανονισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πέτρες, σαν Πρόεδρος και τώρα εξ των Πρασίνων ο κύριος Μίσπο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την ε, Επίτροπο για τη δέσμευση που εξέφρασε για την ε, απανθρακοποίηση των ενεργειακών συστημάτων. Εγώ ανησυχώ για την ταχύτητα της αλλαγής αυτής. Αυτό συζητάμε σήμερα. Αποταχτήκαμε στο Κοινοβούλιο μια δήλωση για το κατεπήγον της αλλαγής του κλίματος και είπαμε ότι θα πρέπει να αξιολογηθούν διάφορες προτάσεις και θα πρέπει να συνάδουν με τις δεσμεύσεις μας σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία του Παρισιού για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμό. Δεν θέλουμε λοιπόν να διακυβεύσουμε το στόχο αυτό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Μα υποσχεθήκατε να ξανακοιτάξετε τον κανονισμό το επόμενο έτος. Αυτό φυσικά μας ικανοποιεί, αλλά δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε άλλη μια λίστα σαν τη σημερινή. Ακόμα και τη σημερινή πρέπει να την κοιτάξουμε. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε ενεργειακές λύσεις που φέρνουν ε, ένα βιώσιμο μέλλον και θέσει απασχόληση για όλου και για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει να μπορούν να επενδύουν σε μελλοντικέ τεχνολογίε. Αν ε, λοιπόν καταλήξουμε με τέτοιου πόρου παροχημένου, τελικά θα καταλήξουμε να έχουμε επενδύσεις οι οποίες δεν θα μπορούν να διατηρηθούν σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, όχι μόνο από πλευρά του περιβάλλοντο. Θα θέλαμε λοιπόν έναν κατάλογο PCI που θα επικεντρωθεί σε ε, δίκτυα ηλεκτρικού και βιώσιμες λύσεις. Να δούμε πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Περίπου 0,5% ε, είμαστε σε ανανεώσιμες μάλλον στο 30% είμαστε σε ανανεμόσιμε ε, ε, πηγές ενέργειας. Το 2050 θέλουμε 80% και μπορεί να υπάρχει ακόμα ε, κάποιο ποσοστό ορεικτών. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε προτεραιότητέ και να δούμε ό,τι αέριο επιτρέπεται θα, πρέπει, επιτρέπεται, θα πρέπει να είναι αέριο πράσινο, όχι από ρηκτά καύσιμα. Και για τις υποδομές θεωρώ ότι χρειάζεται μια αλλαγή προτύπων. Ερώτηση λοιπόν από πλευρά των πρασίνων. Θα κάνετε τον κανονισμό, θα τον επιταχύνετε προκειμένου να κοιτάξουμε στα πλαίσια του επόμενου κανονισμού την επόμενη ρύθμιση, γιατί αυτό θεωρώ ότι θα συνάδει με τι δεσμεύσει που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρο, και να περάσω στην ομάδα των, του ID. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ, Επίτροπε. Καλώ ήρθατε. Καλή επιτυχία στη δουλειά σα. Σα ευχόμαστε να είναι εποφελή ε, η εργασία σα για τα επόμενα χρόνια. Πριν από τις ερωτήσεις, θα ήθελα να εκφράσω κάποιους ε, προβληματισμούς εν είδη αγωγής. Είναι μια συνάντηση σε μια πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή, λίγες μέρες πριν την παρουσίαση της Νέας Πράσινης Συμφωνίας. Μιλώντας με επιχειρηματίες, με διάφορες οργανώσεις, με συνδικάτα, με απλούς πολίτες, ε, συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν Υπάρχει πολύ περιέργεια από πλευρά του και πολλέ προσδοκίε και ανησυχίε όμω παράλληλα. Γιατί φοβούνται ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να πάει πολύ γρήγορα σε σχέση με τις δυνατότητε που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ελπίζω όμως ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πιο ξεκάθαρες ιδέες και εν πάση περιπτώσει θα μου δοθούν επιχειρήματα για να ανασκευάσω λιγάκι ε, τις κινδυνολογίες και τους φόβους. Α πάμε στα δικά μας όμως, τα σημερινά. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντο είναι εκ των κάνεθ για να συμπληρώσουμε την, ε, μια συνδεδεμένη αγορά. Για τον τέταρτο κατάλογο τώρα ήταν αυτά. Για την πέμπτη λίστα ελπίζουμε να υπάρχει μια αποτελεσματική συνεργασία και ένα συνεχίσει διάλογος ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Μια σκέψη για το φυσικό αέριο. Η προβλέψεις για τις ανάγκες, παραδείγματο χάρη η Ιταλία είναι τρίτη η πυρωτική αγορά, μέχρι το 2030 θα είναι κάτω από τα 70 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Και μετά θα πάει από το 2035 στα 69 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Εξακολουθεί να μας απασχολεί αυτό το θέμα σε εθνικό επίπεδο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα στοιχεία, αυτά τα νούμερα ότι πρέπει να τα λάβετε υπόψη στο διάλογό μας. Θα ήθελα να σας αναφέρω και μία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2018 που αναφέρει μία μελέτη όπου μία έξυπνη χρήση του ανανεώσιμου μεθανίου και του έξυπνου υδρογόνου θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε εξοικονόμηση μέχρι το 2050 217 δισεκατομμυρίων. Η ενεργειακή μετάβαση λοιπόν πρέπει να γίνει με προσοχή, πρέπει να τη διαχειριστούμε προσεκτικά. Δεν πρέπει να τη δούμε σαν απειλή, αλλά ως ευκαιρία. Από τη μία δηλαδή θα έχουμε ευκαιρίες για το περιβάλλον, αλλά γιατί όχι και σε επίπεδο θέσεων απασχόλησης. Αυτά έχω να σας πω, δεν είχα συγκεκριμένα ερωτήματα, αλλά ήθελα να σας πω αυτούς τους προβληματισμούς. Ευχαριστώ. Eh, Σας ευχαριστώ εξ ονόματος του ΣΥΑΡΑ, ο κύριος Φανανόρδεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σε μια θέση όπου κατά πάσα πιθανότητα θα αποχωρήσει Brexit. Η συμφωνία αποχώρησης ε, συμπεριλαμβάνει και κάποια ε, εμπλοκή και συμμετοχή σε ό,τι αφορά το κατάλογο PCI μέχρι το 2020 και στη συνέχεια ε, για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Έχουμε δει λοιπόν την τέταρτο κατάλογο PCI που συμφωνηθήκε από τα κρατημέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καταλαβαίνω ότι άλλαξε η επικέντρωση και δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ε, ενοποίηση και την ενσωματώση των ανανεώσιμων και την ε, βιώσιμη προμήθεια, παροχή. Να μας πει λίγο παραπάνω λόγια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ακριβή κριτήρια. Γιατί κάποια έργα ε, βγήκαν από τον κατάλογο. Ένα παράδειγμα, για παράδειγμα, να σας πω το project ε, το γαλλοβρετανικό Aquin για να καταστούν οι αγορές οι ενέργειας πιο αποτελεσματικές με μηδενικές ε, εκπομπές και με ασφάλεια εφοδιασμού και με την αύξηση του ρόλου της ε, ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Είχε περάσει στον κατάλογο PCI, είχε περάσει από τον τεχνικό έλεγχο, αλλά παραλήφθηκε, απορρίφθηκε στην ε, πράξη κατά εξουσιοδότηση. Αναρωτιέμαι, ήταν κατά λάθο αυτή η παράληψη. Και φυσικά έχω και άλλα παραδείγματα τέτοια να δώσω. Αναρωτιέμαι, τι βήματα μπορούν να γίνουν τώρα για να διορθωθούν τέτοιε περιπτώσεις και να συμπεριληφθούν ε, τέτοιες, τέτοια έργα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φανόρντεν. Από τους μία ο κύριος Κοράου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καλημέρα. Καλώ ήρθατε, κυρία Επίτροπε. Χάρηκα που άκουσα τι νέε πράσινε προτάσει και δεσμεύσει ε, τη Επιτροπή να αντιμετωπίσουμε αυτό το παγκόσμιο βάρο στον πλανήτη. Θέλω όμως πρωτού ε, το ε, κραυγάσω να δω συγκεκριμένη πρόεδρο. Υπάρχουν αντιαφισβήτητα θετικά στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ότι θα σταματήσει να, να χρηματοδοτεί έργα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ρεκτά καύσιμα, έστω και από το 2021. Περιμένουμε και μια θετική απάντηση σε ό,τι αφορά το τελευταίο ταμείο μετάβαση, το οποίο ελπίζω ότι θα παραταθεί. Όχι μόνο για τη μείωση της, του του άνθρακα, αλλά πρόσφατα, στην πρόσφατη λίστα, τα project που περιλαμβάνονται είναι πολύ ασαφή. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία. Το Κοινοβούλιο έλαβε την λίστα τελευταία στιγμή. Παρά το γεγονό ότι ήθελε να συμμετέχει πιο πολύ για τον καθορισμό των ορισμών. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, όντω οι εμπειρογνώμονε εξηγούν ότι, ότι μπορεί να έχουν μειωθεί τα project που έχουν να κάνουν με το αέριο, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την χρηματοδότηση. Κατά τρίτον, η χρονική συγκυρία. Υπάρχουν κάποια project τα οποία ακόμα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση τη ΕΤΕΠ. Άρα ο κατάλογο δεν φαίνεται να συνάδει με τι πράσινε υποσχέσεις τη Προέδρου Φάντερ Λάιεν σε ό,τι αφορά την ε, κατάργηση του άνθρακα μέχρι το 2050 και τη Συμφωνία του Παρίσιου. Όλες αυτές λοιπόν οι διαφορές υπάρχουν. Επειδή είναι πράξη κατά το κοινοβούλιο μπορεί να πει ένα ναι ή ένα όχι για το σύνολο της πρότασης. Τι θα γίνει λοιπόν αν απορριφθεί η πρόταση, για εξηγήστε μας. Θα κοιτάξουμε ένα τρίτο κατάλογο, ο οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ΕΤΕΠ. Και επίση μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι τα project τα οποία έχουν να κάνουν με το αέριο θα μπορέσουν να χρηματοδοτούνται από το τρέχον και το θεμαρατικό CEF. Θέλω συγκεκριμένες δεσμεύσεις για να αλλάξουν και οι διαδικασίες για την επιλογή των προγραμμάτων, αλλά και τα ίδια τα προγράμματα στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση από την ΚΟΕ, η κυρία Έρνστ, η οποία είναι στη θέση εδώ της κυρίας Ματίας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να παρουσιάσω την απόψη της ομάδας μας. Νομίζω ότι στο σύνολό του, στο σύνολό τους, τα project, τα έργα, διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προαγάγει ακριβούς αγωγούς αερίου και, για παράδειγμα, με το Αζερβαϊτζάν. Αυτές οι υποδομές ε, δεν θα μπορέσουν ποτέ να χρησιμοποιηθούν για το πράσινο αέριο. Ποτέ. Αυτό μας ανησυχεί. Ότι και πάλι χάνουμε μια ευκαιρία. Χάνουμε μια ευκαιρία για να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τις ανανεώσιμες. Αυτό μας λυπεί. Τα έργα υδρογόνου, τα οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ενέργεια, δεν υπάρχουν καν στον κατάλογο. Μα πού ζούμε ο κανονισμός TEN-E ε, προκειμένου να προωθηθούν αυτά τα προγράμματα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια αλλαγή στα κράτη-μέλη για να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή προκειμένου να έχουμε πραγματικά ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Το αέριο, από ό,τι μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι κάτι μεταβατικό. Αυτό πραγματικά είναι ένα περίεργο α, συμπέρασμα. Δεν είναι μεταβατική τεχνολογία, αν προγραμματίζουμε τόσα λεφτά και τόσα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν κλείνει τα μάτια. Εστρατιφλή σε ό,τι αφορά και το μεθάνιο. Αυτό είναι εξαιρετικά επιβλαβές ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποδομή για το αέριο είναι επαρκής, επαρκέστατη αυτή που υπάρχει τώρα σε ό,τι αφορά τις ανάγκες αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναρωτιέμαι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δαπανά πόρους και θέλει να δαπανήσει περαιτέρω πόρους προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης έχουμε 55 έργα άνθρακα. Είναι πραγματικό σκάνδαλο αυτό και δεν συνάδει με τη Συμφωνία του Παρισιού. Επικρίνουμε λοιπόν το γεγονό αυτό και λέμε δημόσια ότι είναι λάθος το βήμα αυτό. Δεν με νοιάζει Ποιο θέλει, τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμένα αυτό που με νοιάζει και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι βγάζουμε δεδυράμβους και τελικά αποφασίζουμε για μία λίστα η οποία είναι εντελώς απαράδεκτη. Σκανδαλώδης θα έλεγα. Thank you very much. So with this we are... Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι ολοκληρώσαμε τον ε, πρώτο γύρο. Πολλές οι ερωτήσεις, πολλές οι προτάσεις. Περνάμε στο δεύτερο γύρο. Έχω 15 συναδέρφους που έχουν ζητήσει το λόγο στο δεύτερο γύρο και προτείνω να κλείσουμε το κατάλογο αν συμφωνείτε όλοι. Γιατί αλλιώ θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Α, εσά σα έχω στο κατάλογο, ναι. Ωραία. Εσεί τώρα να απαντήσετε στου συντονιστέ καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Εσείς κύριε Λένερτς, με την ερώτησή σας θέσατε τις βασικές αρχές. Το θέμα της ασφάλειας και του εφοδιασμού είναι πολύ σημαντικά σε ικανοποιητικέ τιμές. Και το βλέπετε και από τον τέταρτο κατάλογο προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Υπάρχουν και προγράμματα που ξεκίνησαν με προηγούμενους τέτοιους καταλόγους και συνεχίζονται σε περιοχές που ανησυχούν για την διασυνδεσιμότητά τους και για την ασφάλεια εφοδιασμού. Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε την συνδεσιμότητα. Παντού υπάρχουν ε, τερματικά υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τώρα, κάποιοι από εσά. Με ρώτησαν και εξέφρασαν ε, απόψεις για νέα προγράμματα. για το ρόλο των ε, αυτοκινήτων κατά την μετάβαση. Σήμερα το φυσικό αέριο είναι το τέταρτο στο ενεργειακό μας μείγμα. Και είναι αλήθεια ότι ένα μεγάλο μέρος εισάγεται. Στον τέταρτο κατάλογο okay, βλέπουμε 32 προγράμματα φυσικού αερίου που αντιμετωπίζουν ακριβώς αυτό το θέμα των υποδομών χρειάζεται διαφοροποίηση και ασφάλεια εφοδιασμού. Και είναι σαφές ότι αν ε, στρεφόμαστε προς το μέλλον, το 2050 θέλουμε να έχουμε ουδετερότητα όσον αφορά το φυσικό αέριο. Και γι' αυτό πρέπει και να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση και αναθεώρηση του κανονισμού διαγωνισμών πρώτα απ' όλα βάσει των προτεραιοτήτων μας έτσι ώστε να είμαστε δέτεροι το 2050. πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ε, νέες τεχνολογίες. Τα κριτήρια επιλογής τώρα για τους καταλόγους κοινών προγραμμάτων περνάνε από την διαδικασία βέβαια λήψης ε, αποφάσεων και περνάνε και από τη διαδικασία ρογής. Και τα περισσότερα περνάνε από σε βάθος αξιολόγηση πριν να αποφασίσει για μια πρωτοβουλία επιτροπή. Το ερώτημα για το τι αποτελεί τη βάση της αναθεώρησης που απαιτείται για τον σημερινό ε, κατάλογο, η αναθεώρηση γίνεται κάθε δύο χρόνια. Και ως αποτέλεσμα η πέμπτη, ο πέμπτος κατάλογος θα αναθεωρηθεί το 2021. Ε, πρόκειται για μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Και χρειάζεται χρόνος βέβαια για την κατάρτιση του καταλόγου. Πολύ χρόνος. Έχει ήδη ξεκινήσει βέβαια η δουλειά με το σημερινό τεχνικό πλαίσιο. Όπως όμως είπα, Ακόμα και με το σημερινό πλαίσιο μπορούμε να κάνουμε πολλά και σκοπεύω να κάνω πολλά. Πρώτα απ' όλα, είναι σημαντικό να γίνεται η αξιολόγηση βιωσιμότητας των προγραμμάτων Ευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας. Και τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ενισχυμένους ελέγχους. Αλλά όχι μόνο να δούμε είναι ε, το πρόγραμμα χρήσιμο. Επίσης, πρέπει να αξιολογούμε και τις επιπτώσεις των αντίκτυπων όσον αφορά τα αίρια του θερμοκηπίου. Και να λάβουμε υπόψη μας και τις επιδόσεις των υποδομών για να δούμε πόσο ρηπαίνουν. Uh, um, Οπότε αυτή είναι η απάντηση. Ο, το φυσικό αέριο πρέπει να παραμείνει ως εργαλείο για την μετάβαση Φυσικά θα υπάρχει και αναθεώρηση εφόσον έχουμε και το βιοαέριο και υδρογόνο κλπ. Υπήρξαν ερωτήσεις για τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από όσο γνωρίζω, η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας έρχεται για να ενημερώνει την Επιτροπή σας. Εβδομάδες ε, ήρθε εξάλλου πριν παρουσιάσει τον κατάλογο ε, και ο κύριος Αρίας Κανιέτε και προηγουμένως υπήρχαν συναντήσεις και υπήρξε διαφάνεια. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι μια δικασία από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή τα προγράμματα ετοιμάζονται από τις χώρες ε, μέλη Υπάρχει ομάδα εμπειρογνωμόνων επίσης, ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων που τα αξιολογεί σε συναντήσεις. Και πρέπει να υπάρχει συνένεση για τα προγράμματα. Αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Και είμαι έτοιμη να παρουσιάσω εδώ στην Επιτροπή Ήτρε τα διάφορα στάδια της διαδικασίας και ποια είναι αυτά τα στάδια κλειδί της διαδικασίας. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των υποδομών αναλύεται κατά πόσο χρειάζονται πρώτα απ' όλα τα υποψήφια προγράμματα ή όχι. Και αυτό θα γίνει εν ώψη του 2021. Πριν ληφθεί απόφαση η οποία θα ληφθεί στα μέση του 2021. Είπαμε ότι κάθε δύο χρόνια θα ετοιμάζεται νέος κατάλογος προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Αναφέρθηκα και στις ε, ομάδες εργασίας και υπάρχουν και περιφερειακές ομάδες εργασίας. όπως των Βαλτικών χωρών, ε, της Βόρειας Θάλασσας, ε, συνεργασία ε, Βόρεια-Νότια Ευρώπη, συνδεσιμότητα. Υπάρχουν συναντήσεις για τα προγράμματα και θα φροντίσω να προσκληθούν και μέλη της Επιτροπής σας. Σε αυτές τις συναντήσεις υψηλού επίπεδου ομάδων εργασίας. Ο κύριος Γκονζάλης τώρα με ρώτησε πολύ συγκεκριμένα ποια είναι η ισορροπία ανάμεσα στα διάφορα προγράμματα ηλεκτρισμού. Όπως βλέπετε στο νέο κατάλογο, τον τέταρτο, υπάρχουν λιγότερα προγράμματα φυσικού αερίου από ό,τι προηγουμένως. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι δεν πρόκειται για αγγίση, πρόκειται για μια εκ των προτέρων προϋπόθεση. Κάποια από τα προγράμματα που ήταν στον τρίτο κατάλογο βλέπετε ότι δεν είναι πια στον τέταρτο. Ακριβώς αφαιρέθηκαν γιατί δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Με ρωτήσατε επίσης συγκεκριμένα με το πρόγραμμα Aquint που περιλαμβάνεται και αξιολογήθηκε από την Περιφερειακή Ομάδα θετικά. Αλλά όπως είπα, στη συνάντηση υπήρχαν τέσσερις υποψήφοι ε, για τη στεσιμότητα Γαλλίας Ηνωμένου Βασιλείου. SB, ε, Και υπάρχει η περίπτωση να υπάρχει παραπάνω προσφορά από όσο χρειάζεται. Και η Γαλλία δεν θέλει το Aquint να υπάρχει πια στον κατάλογο Και αυτή είναι μια προϋπόθεση ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να στηρίξουν τον κατάλογο. Θέλω επίσης να σας μιλήσω για την δανειακή πολιτική IPL. Όπως γνωρίζετε, πριν από δύο εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έκανε την ανακοίνωση για την ε, πολιτική της δανεισμού ότι θα είναι διαφορετική και θα ευθυγραμμίσει τις δραστηριότητες της προς την Συμφωνία του Παρισιού. Αλλά οι επενδύσεις σε προγράμματα φυσικού αερίου και στα πλαίσια του πολιτισμού οικονομικού πλαισίου είναι ακόμα επιλέξιμα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λοιπόν υιοθέτησε νέες κατευθυντήριες γραμμές για την χρηματοδότηση επενδύσεων όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να ξέρουμε δηλαδή ότι μπορεί ακόμα να εγκρίνει χρηματοδοτήσεις η ΕΕΠ για δάνεια σε προγράμματα όπου ενέχεται το φυσικό αέριο εφόσον έχουν ήδη τεθεί ως υποψήφια τα προγράμματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις. Περνάμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων τώρα. Όπως είπαμε έχουμε 15 συναδέρφους, γι' αυτό σας παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας. Ένα λεπτό καθένας για ερώτηση. Για τελειώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τηρήσουμε το χρόνο μας. Η κυρία Καρβάλιο είναι η πρώτη που έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε. Σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια έργα που δεν συμπεριλαμβάνονται στον τέταρτο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος ΕΚΕ. Μιλάω για έργα που αφορούν την Ιβυρική Χερσόνησο και την διασυνεση Ισπανίας, Πορτογαλίας, Γαλλίας. Θα ξέρετε ίσως ότι έγινε μια σύνοδος τον Ιούνιο του 2018 όπου ε, οι επικεφαλείς της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας αποφάσισαν να προωθήσουν τη διαλειτουργικότητα των τριών και διασύνδεση αυτών των τριών χωρών. Είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια του ανεφοδιασμού και την ε, δυνατότητα διαφορετικής ε, προμήθειας διαφορών δρόμων ανεφοδιασμού σε ενέργεια για την Ιβυρική Χερσόνησο. Μιλάω για την πρώτη διασύνδεση Ισπανίας-Πορτογαλίας ε, και μία άλλη ε, στα νοτιοανατολικά, στα σύνορα ε, Γαλλίας-Ισπανίας. Ε, Θα είναι πολύ σημαντικό για την Ιβηρική Χερσόνησο, την ασφάλεια των εφοδιασμού και την βιωσιμότητα ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί αυτά τα έργα δεν τα συμπεριλάβατε γιατί δεν τα θεωρήσατε αξιοσημείωτα. Ευχαριστούμε κύριε Καρβάλιο. Ο κύριος Μπούζεκ. Αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω ότι μητρική μου. Τα πορτογαλικά. Ευχαριστώ Επίτροπε. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε για πρώτη φορά στην Επιτροπή μας. Δεν είναι πλέον μία ακρόαση, είναι μία σοβαρή συζήτηση. Πάντα σωστή, καλό πράγμα είναι να κάνουμε τέτοιες ε, συζητήσεις για τα ΕΚΕ. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να μας ικανοποιήσει σε όλες τις προσδοκίες μας. Θα ήθελα και εγώ να παραπονεθώ για δύο-τρία έργα, τα οποία έβρισκα αρκετά σημαντικά. Θα ήθελα παρόλα αυτά, καταρχάς να μιλήσω για κάτι πιο σημαντικό, κάτι πιο γενικό. Αυτός ο κατάλογος συζητιέται επί μακρόν. Καλό είναι αυτό. Γιατί παλιά συζητήσαμε τον τέταρτο ε, κατάλογο. Ε, ο διευθυντής της Γενικής σας Διεύθυνσης ήταν ε, και παρόν, είχε έρθει εδώ και το συζητήσαμε το θέμα αυτό με το κοινό. Το συζήτησε δηλαδή η Κομισιόν με το Κοινοβούλιο. Ας συνεχίσουμε σε αυτόν τον ρυθμό. Ας κάνουμε αυτές τις ζητές συζητήσεις μέσα σε ένα-δυο μήνες. Είναι μια αρκετά σωστή αλλαγή πολιτικής. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και τις διασυνδέσεις σε επίπεδο ηλεκτρικής ενέργειας για μας είναι πολύ σημαντικό. Ειδικά όταν συζητούσαμε τον τρίτο κατάλογο, το απαιτούσαμε αυτό. Η κατεύθυνση είναι σωστή. Και όπως είπατε κι εσείς, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ένα σημείο αφετηρίας για οτιδήποτε κι αν κάνουμε. Οι διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικές, η βιωσιμότητα είναι πολύ σημαντικές, η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική, όπως ανέφερε και ο κύριος Έλα, ο κύριος Έλερ, συγγνώμη, και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δίκτυα για βιοαέριο, για συνθετικό αέριο και όχι μόνο για την μεταφορά φυσικού αερίου. Θα πρέπει να περάσουμε και στο υδρογόνο επίσης. Θα πρέπει να ετοιμαστούμε και σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες και τη συζητάμε ήδη στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ. Σε δύο χρόνια θα έχουμε αυτή την οδηγία που είναι πολύ σημαντική για την Επιτροπή μας. Ο επόμενος ομιλητής. Κυρία Καρφίν, ευχαριστώ που ήρθατε εδώ, Επίτροπε. Η ενέργεια δεν είναι ένα αγαθό, ε, βασικό αγαθό, είναι ένα βασικό κοινωνικό δικαίωμα. Έχουμε 80 εκατομμύρια πολίτες σε όλη την Ευρώπη που έχουν ενεργειακή φτώχεια και επιλέγουν ε, αν θα φάνε ή αν θα ζεσταθούν ή αν θα δροσιστούν. Χρειαζόμαστε ε, ταχαίως αναθεώρηση ε, των ε, διευρωπαϊκών δικτύων. Έχουμε 32 ε, ε, έργα φυσικού αερίου και 6 αέρια πετρελαίου σε αυτό το κατάλογο. Πώς μπορώ να το υπερασπιστώ αυτό απέναντι στην κόρη μου που θέλει να σώσει τον πλανήτη όπως όλοι οι νέοι. Θέλουμε η Ευρώπη να δίνει το παράδειγμα στη νέα πράσινη επανάσταση. Να υπάρχουν νέες πράσινες ε, θέσεις απασχόλησης για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Σε ό,τι αφορά την μετάβαση, είδα την ε, επέκταση του καταλόγου δεν πρέπει να μιλάμε ως για πολιτική, Πρόεδρε. Μιλάμε, πρέπει να μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης. Και ε, η Ευρώπη να παίξει ηγετικό ρόλο στη Νέα Πράσινη Συμφωνία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, με βρώμικα έργα φυσικών ε, καυσίμων. Θα πρέπει να υλοποιήσουμε την Πράσινη Συμφωνία, θα πρέπει να δώσουμε δουλειά σε όλα τα νέα κορίτσια στο μέλλον. Και πραγματικά είμαι θλιμμένη που ενδεχομένως το Ηνωμένο Βασίλειο θα φύγει από την Ευρώπη, αλλά πρέπει να ηγηθούμε στη νέα πράσινη μετάβαση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια διαδικασία. Πρέπει να είμαστε ηγέτες στην πολιτική. Πρέπει εδώ να σε τιμήσω Τζέρζι, Μπούζεκ και το Μιγγέλ. Γιατί στην αρχική ε, ακρόαση εγώ του έφερα αντιρρήσεις. Ε, αυτός όμως μας έδειξε το παράδειγμα για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Μίλησε με πολύ σημαντικά λόγια για την ενεργειακή φτώχεια και ελπίζω στη, στο μέλλον να δώσετε αυτό το παράδειγμα για όλες τις μελλοντικές γενιές. Επίτροπε. Ο κύριος Ζωρίνιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, εδώ είμαι. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ για τη νέα σας εντολή, για το νέο σας αξίωμα. Ελπίζω να συνεργαστούμε καλά. Επί πολλά χρόνια η Κομισιόν δούλεψε με την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία για να ενισχύσει την διασυνδεσιμότητα ανάμεσα στις τρεις αυτές χώρες, στον τομέα του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση τις διατάξεις ε, του κανονισμού για την ενέργεια. Υπάρχουν μεγάλες ε, κυβερνητικές δεσμεύσεις ανάμεσα στις τρεις χώρες, χώρες για να προωθηθεί αυτή η συμφωνία. Κι όμως, με κατάπληξη βλέπω, υπάρχει κάτι το αρνητικό. Ε, δόθηκε αρνητική ε, γνωμοδότηση για την κατασκευή του αγωγού του Σινές στην Πορτογαλία. Και επίσης Ακούσαμε σήμερα ότι ένας αγωγός αερίου δεν μεταφέρει μόνο αέριο από φυσικά από καύσιμα, αλλά και καθαρό αέριο. Πιστεύετε ότι ο στρατηγικός στόχος του, της ποικιλομορφία των φυσικών πηγών ενέργειας πρέπει να λυθεί υπόψη και να χρηματοδοτούμε τέτοιου είδους έργα, λαμβάνοντας υπόψη το στοιχείο της ε, συνδεσιμότητας και διαλειτουργικότητας. Επίσης μπορείτε να παρακάμψετε την άποψη κάποιων ρυθμιστικών αρχών, γιατί υπάρχουν που συμφωνούν ε, με κάποια έργα και θα υποφεληθεί η κοινωνία τους. Πώς ε, μπορούμε να αποφύγουμε ε, συγκυριακές βραχυπρόθεσμες αποφάσεις να μας διαιρέσουν στα θέματα της ενέργειας μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Madame Judith Banding. Sorry. Thank Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ σήμερα, Κάντρα, για να μας μιλήσετε για τους διασυνδεσιμότητα. Χάρηκα που στην αρχή της παρουσίασής σας ε, μας επιβεβαιώσατε ότι η περίοδος ελέγχου για την ε, έλεγχο της ε, λίστας αυτής ε, παρατάθηκε για κάποιους μήνες γιατί δεν έχει όμως νόημα να τον εξετάσουμε τον κατάλογο αυτό, αν δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγή. Άρα, πρώτη ερώτηση, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι είστε ε, ανοιχτοί να αναθεωρήσετε αυτό τον τέταρτο κατάλογο PCI. όπως και πολλοί φίλοι εδώ, δεδομένη και τη έκτακτη κατάσταση για το κλίμα στο Green Deal, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι απορρίπτονται οποιαδήποτε τέτοιοι διασύνδετες. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να απορρίψουμε τίποτα τέτοιο. Δεν μπορούμε να απορρίπτουμε τέτοιες υποδομές οι οποίες τεχνικώς είναι κατάλληλες. Η σύνδεση μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας, για παράδειγμα, θα αμα, ωφελούσε τους παρόχους ενέργειας και θα υποστήριζε επίσης την ανανεώνηση των, την ανανέωση των σχεδίων στην ε, Νοτιοανατολική Αγγλία. Και οι δυνατότητες ε, όλων των υποδομών που προτείνονται είναι πολύ χαμηλότερα από τις ε, απαιτήσει που υπάρχουν και τις προδιαγραφές που υπάρχουν για τόσο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Άρα η απόρριψη αυτών και η απόρριψη όλων των άρτιων τεχνικών υποδομών, θέλω να μου υποσχεθείτε ότι θα αναθεωρηθεί δεδομένη τη περίοδου α, χάρτος που δίνεται και τη σημασία τη Πράσινη Συμφωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπλό από του Πράσινου. Καλημέρα και αντικαθιστώ τον κύριο Μπλό, ε, κυρία Πρόεδρε, Επιτροπέ αναλάβατε τα καθήκοντά σας μαζί και εμάς και γνωρίζετε ότι μεγάλη ευθύνη φέρουμε γιατί από εμά και από τις αποφάσεις μας εξαρτάται να εξασφαλίσουμε το κοινό μας μέλλον. Στην COP21 λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίναμε μάλλον για την ε, προηγούμενη εβδομάδα ένα ψήφισμα σε ό,τι αφορά το μέλλον του περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Εμεί, λοιπόν ε, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνουμε αποφάσει που θα είναι καθοριστικέ μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα γιατί τα έργα αυτά θα καθορίσουν ε, τι εκπομπέ του διοξιδίου του ανθρακά. Σήμερα όμω βασιζόμαστε σε ένα κανονισμό ΔΕΔΕ του 2013 σε ό,τι αφορά Τη ε, δεσμεύση τη Ευρώπη στην Παρίσι, θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε στο ύψο των περιστάσεων, όπω είπαν και οι συνάδελφοι. Θα πρέπει να υλοποιηθεί ο κανονισμός βέβαια, Μας μιλήσατε για τις ε, προηγούμενες λίστες. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί παταγώδη αποτυχία σε ό,τι αφορά τα έργα τα οποία είναι κατάλληλα. Θα πρέπει να πάρουμε λοιπόν να δείξουμε την τόλμη και πολιτικό θάρρος για να βάλουμε ένα στόπ στα έργα αυτά και από σήμερα να ξεκινήσουμε σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρασταντεύσκη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Επιτρέπε, μια ερώτηση να κάνω. Ποιες θα είναι οι συνέπειες και αυτό είναι σημαντικό για μας, αν επανέλθουμε από την τέταρτη λίστα στην τρίτη. Επειδή δεν θα γίνει αποδεκτή η τέταρτη λίστα. Περιλαμβάνονται κάποια στρατηγικά προγράμματα κλειδί. Να εντοπίσω ένα και μόνο τον αγωγό τη Βαλτική. Ένα πάρα πολύ σημαντικό σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος για την Κεντρική Ευρώπη. Ενδεχομένως να μην το γνωρίζετε, αλλά τον Νοέμβριο η Πολωνία, η χώρα μου, ενημέρωσε την Gazprom, την οποία φαντάζομαι θα ξέρετε, ότι η σύμβαση Γιάμαλ θα εκπνεύσει στα τέλη του 2022. Και κατά 80% εξαρτώμαστε από ρωσικές ε, προμήθειες. Αυτός ο όγκος θα αντικατασταθεί από εισαγωγές από άλλες πηγές συμπεριλαμβανομένου και του αγωγού της Βαλτικής στον, στη λίστα 4. Αυτά τα προγράμματα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά για το περιβάλλον. Γιατί θα μειώσει τα σωματίδια κατά 54% καθώς και το διοξείδιο του άνθρακα. Ρωτώ λοιπόν, δεν πιστεύετε κάποια ρεζοσπαστικά ε, αλλαγέ ό,τι αφορά το περιβάλλον ε, μπορεί να έχουν αντιπαραγωγικό αποτέλεσμα. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Σα παρακαλώ να είστε σύντομοι, γιατί έχουμε 15 λεπτά παραπάνω, αλλά να είστε παρακαλώ αυτά σύντομοι. Κυρία Νίπλερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και την Επίτροπο που είναι διατεθειμένη να κάνει αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ξεκινήσατε λέγοντα, Επίτροπε, ότι υπάρχει αυτό ο φιλόδοξο στόχο για την ε, περιβαλλοντική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Θεωρώ ότι τεχνολογικά είναι δυνατό αυτό και θα πρέπει να είναι και οικονομικά επιτεύξιμο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω από πού θα έρθει όλο αυτό το ηλεκτρικό που χρειαζόμαστε για να είμαστε περιβαλλοντικά ουδέτεροι και πώς θα καταφέρουμε να είναι λογικές και οι τιμές του ηλεκτρικού στο μέλλον. Εγώ είμαι από τη Βαυαρία και έχουμε παραγωγική βιομηχανία στην ε, περιοχή μου. Κοιτάω για παράδειγμα την χημική βιομηχανία. Τι χρειαζόμαστε για κατανάλωση ρεύματος. Μέχρι το 2050 θα δεκαπλασιαστούν οι ανάγκες μας. Πώς θα καλύψουμε λοιπόν ε, αυτές τις ανάγκες. Πώς θα καλυφθούν ε, αυτές οι κλίμακες που θα χρειαστεί για παράδειγμα να καλύπτονται πολύ μεγαλύτερες ανάγκες, γιγαντιές ε, πραγματικά διαφορές. Θα ήθελα λοιπόν μια απάντηση και να σας παρακαλέσω να μου πείτε από πού θα έρθει το ηλεκτρικό αυτό. Θα πρέπει να φροντίσουμε να μπορούμε να το καταβάλουμε. Θα ήθελα λοιπόν επίσης να υποστηρίξω τον συνάδελφο κύριο Πέτερσον. Δεν θέλουμε μόνο α, αξιολογήσεις βιωσιμότητας, αλλά πλήρης μελέτης αντικτύπου για το πώς ε, τα πετύχουμε όλα αυτά, όπως γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βάης. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε. Είπατε ότι θέλετε να βάλετε τον κόσμο στο κέντρο. Το εκτιμώ ιδιαίτερος. Υποθέτω εννοείται και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπη. έτσι. Σήμερα μιλάμε για την διασυνδεσιμότητα και για τις υποδομές πολύ σημαντικά κομμάτια του παζλ. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω για τις ψηφιακές λύσεις και τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε την Ενεργειακή Ένωση ως φιλοδοξία, αλλά να είμαστε και δυνατοί σε ψηφιακέ λύσεις. Οπότε ανάμεσα στι ψηφιακές λύσεις και την ενέργεια δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια γέφυρα. Δεν θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει μια πλατφόρμα ώστε η τεχνολογία να επιτρέπει η ενέργεια να κυκλοφορεί ελεύθερα με ανανεώσιμες, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έτσι να αυξηθεί η ποσότητα της ενέργειας που θα κυκλοφορεί και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που πρέπει να έχουν την καλύτερη τιμή για την ενέργεια. Θέλω τη σκέψη σας πάνω σε αυτά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κάφε από τους Πρασίνους, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο κυρία Σίμψον. Πιστεύω κι εγώ ότι το θέμα της πρόσβασης ενέργειας σε καλές τιμές είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν πρέπει να αφήνουμε στην πάντα βέβαια το θέμα των εκπομπών. Είπατε ότι δεν θέλετε προγράμματα τα οποία δεν συμμορφώνονται με το Παρίσι. Δεν μπορούμε τη μισή θητεία να την περάσουμε χρηματοδοτώντας ε, δεινόσαυρους. Οπότε νομίζω ότι εσείς ακολουθείτε την γραμμή που λέει ναι μεν θέλω να συμμορφωθώ με το Παρίσι αλλά δώστε μου χρόνο. Οπότε το ρώτημα κλειδί είναι μπορούμε να κάνουμε χωρίς φυσικό αέριο. Εγώ πιστεύω πως ναι και όπως είπατε κι εσείς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημοσίευσε έναν χάρτη πορείας της πολύ φιλόδοξο. Οπότε θα πάει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πιο μακριά από εμάς Υπάρχει το πρόγραμμα του Σάνων στην Ιρλανδία για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και φαίνεται ότι ευθυγραμμίζεται και στο πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη ρογμάτωση. Οπότε το δίκτυο φυσικού αερίου θα πρέπει να είναι αυτό που λέμε future proof, που σημαίνει ότι τα διάφορα φυσικά αέρια θα πρέπει να έχουν πολύ μικρό αποτύπωμα. Συνεπώς ρωτάω, ο κατάλογος των προγραμμάτων τελικά θα περιλαμβάνει μόνο βιώσιμα προγράμματα που όντως θα ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της, ε, του Παρισιού. Η κυρία Τόκ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Πολλοί άνθρωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλούν για τον άνθρακα και η Πολωνία ξέρετε ότι είναι μια ιστορική χώρα και ότι ο άνθρακας αποτελεί μέρος της δικιάς μας παράδοσης. Ακούω επίσης από την περιοχή Σελίζια, χτες είχαμε ε, κάποιες ε, εκδηλώσεις και μαζί γιορτάσαμε και είπαμε πόσο σημαντικός είναι ο άνθρακας για τη χαλιβουργία κάτι το οποίο θα συνεχίσει να ισχύει. Ο άνθρακας δεν είναι ε, κάτι κακό. Χρειάζονται έτσι κι αλλιώς οι αγωγοί για την μεταφορά και από τη Σαχάρα του φυσικού αερίου. Οπότε εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στην πράσινη αυτή μετάβαση και από πλευράς ε, των πολωνικών συνδικάτων ε, Solidarity της Ελεγγύης. Θα ήθελα να επαναλάβω όμως αυτό που είπα και πριν, ότι το φυσικό αέριο πρέπει να αποτελεί μέρος του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου σχεδίου ενεργειακής μετάβασης. Η στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ξεκάθαρη. Το θέμα της υλοποίησης όμως δεν μου φαίνεται καθόλου ρεαλιστικό, έτσι όπως παρουσιάζεται από την Επιτροπή. Η μετάβαση αυτή κοστίζει πάρα πολλά χρήματα και δεν είναι και συγκεκριμένη. Κανένας δεν καταλαβαίνει πώς ακριβώς θα γίνει και πόσο θα κοστίσει. Ποιο θα είναι το τίμημα. ο ανθρακάς χρειάζεται και για τη θέρμανση στα νοικοκυριά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κονδύλια για την ε, ανάπτυξη αυτού του είδους ενέργειας στο εσωτερικό της χώρας. Αλλιώς χρειαζόμαστε εναλλακτικέ λύσεις και πραγματικά ε, πρόκειται για δισεκατομμύρια σλότ, σλότης. Οπότε επαναλαμβάνω αυτό που είπε και ο κύριος Έλερ, ότι ναι, ε, ασφάλεια, προσβασιμότητα και σε καλές τιμές, αλλά και στην Πολωνία να ξέρετε ότι χρειαζόμαστε συμβατική ενέργεια. 200 εκατομμύρια ευρώ. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Ε, το μισό χρόνο θα χρησιμοποιήσω εγώ από ό,τι είπε συνάδελφος, από αυτό που χρησιμοποιήσε η συνάδελφος. Ε, θα ξεκινήσω με τα επιχειρήματα του κύριου Έλλερ. Εγώ έρχομαι από μια χώρα, την Ελλάδα, που έθεσε πολύ φιλόδοξους στόχους για να μην περιλαμβάνεται άνθρακα στο ενεργειακό της μείγμα το 2028. Τώρα για το φυσικό αέριο, εσείς στον κατάλογο ε, τον τέταρτο αναφέρεστε στην Καβάλα και στο πρόγραμμα εκεί, όπως επίσης και αυτό της Αλεξανδρούπολης. Εγώ θέλω να ρωτήσω για τον επόμενο κατάλογο, το πέμπτο. Το ερώτημά μου δηλαδή είναι, τα νέα κριτήρια θα έχουν σαν αποτέλεσμα τα δύο αυτά προγράμματα, ε, θα τα συμπεριλάβει στο νέο κατάλογο και αν θα ολοκληρωθεί, θα υλοποιηθεί πλήρως το πρόγραμμα προκειμένου να περάσουμε στη μετάβαση. Ξέρω ότι άλλε χώρες προχωράνε πολύ γρήγορα για να ε, αλλάξουν ε, το δικό τους μείγμα, αλλά καταλαβαίνει το θέμα των υποδομών παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ευχαριστούμε, κυρία Γκινάτοπ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για τη δουλειά που κάνετε όσον αφορά τα προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος. Υπάρχουν υποχρεώσεις συγκεκριμένες για την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή και την πρόκληση αυτή υπεύθυνα. Πρέπει λοιπόν από κοινού να βάλουμε τις προσπάθειές μας για να έχουμε ασφάλεια εφοδιασμού, αλλά να μπορούμε να έχουμε και ενέργεια σε καλές τιμές. Ο τέταρτος κατάλογος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Χαίρομαι λοιπόν που ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει πολλά προγράμματα με ανανεώσιμες πηγές για τον ηλεκτρισμό αλλά και για το φυσικό αέριο. Εφόσον υλοποιηθούν αυτά, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταλήξει να έχει το 2025 ένα πολύ αποτελεσματικό δίκτυο φυσικού αερίου και καθαρό. Οπότε το κόστος και ο κίνδυνος της μετάβασης, κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αν δεν το πετύχουμε αυτό, ε, θα κοστίζει υπερβολικά πολλά χρήματα για τις ενδιαφερόμενες χώρες. Οπότε ρωτάω πώς θα διασφαλίσετε εσείς ότι σε περίπτωση αλλαγής στον τρέχοντα κατάλογο ε, του ΕΚΕ δεν θα ξεχαστεί καμία περιφέρεια. Ευχαριστούμε. Η κυρία Πάουλου, η τελευταία. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Μου αρέσει η απόψή σας με βάση κάποια νούμερα που μας δώσατε. Η Κομισιόν το 2015 είπατε ότι για το μεθάνιο έχουμε απώλεια. Δηλαδή, απώλεια του μεθανίου μέσω των αγωγών και των αντλίων, αντλιών κατά 2,7%. Το μεθάνιο είναι πολύ ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου. 30 φορές ε, πιο ισχυρό από το διοξίδιο του άνθρακα. Και αυτό σε 30 χρόνια. Σε 10 χρόνια, ε, μέσα σε μια δεκαετία, α πούμε, είναι ακόμα πιο ισχυρό. Αν λάβατε υπόψη σε αυτά τα νούμερα, τότε μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα ότι ο άνθρακα ε, παράγει ένα τόνιο, ε, τόνο διοξιδίου, του άνθρακα ε, την ώρα, ενώ τα εγκαταστάσει εγκαταστάσεις ε, από φυσικά ε, καύσιμα 0,6, ενώ το μεθάνιο πολύ περισσότερο. Δηλαδή, αν περάσουμε από το άνθρακα στο φυσικό αέριο, θα έχουμε μεγάλη εξοικονόμηση. Δεν θα μπορέσουμε να σεβαστούμε τα όρια του Παρισιού εάν δεν κάνουμε αυτή τη μετάβαση. Θέλω να μου πείτε την άποψή σα για αυτέ τι εκπομπέ και να σα υπενθυμίσω ότι δεν είναι οι αρχικέ εκπομπέ που γίνονται στο πηγάδι ε, και κατά την μετακίνηση μέσω του αγωγού ας πούμε, στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για τη δέσμευσή σας να εκτιμήσετε τη βιωσιμότητα αυτή. Θα ήθελα να μου πείτε πώς θα εφαρμόσετε τα κριτήρια. Γιατί δεν είναι όλα τα κριτήρια ποσοτικά. Θα τα μεταφράσετε σε δικαιώματα σε διοξείδιο του άνθρακα ή σε δικαιώματα καύση ας πούμε των δασών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα της Γερμανικής Περιβαλλοντικής Υπηρεσίας που είπε ότι ο κόστος ε, ε ενός τόνου διοξίδου του άνθρακα είναι 1080 ε, ευρώ ανά τόνο διοξιδίου του άνθρακα. Αυτά τα νούμερα θα συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση βιωσιμότητας που θα κάνετε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε για την ενέργεια σήμερα και για την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας που χρειαζόμαστε. Στη σημερινή συζήτηση για τις ενεργειακές υποδομές και τα έργα τα σχετικά, διερωτώ με για πολλά πράγματα ε, και θα ήθελα να μου διευκρινίσετε κάποια. Πώς είναι δυνατόν ε, πολλά από τα project ε, να είναι υποδομές φυσικού αερίου ακόμα και σήμερα. Ενώ είναι σαφώ ότι η Ευρώπη πρέπει να ξεκόψει από το φυσικό αέριο. Το είπαν και οι συναδελφοί μου και θέλω να το τονίσω κι εγώ. Παρότι το ποσοστό των ε, έργων μειώθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο κατάλογο, πώ μπορείτε να μα εγγυηθείτε τώρα, Κομισιόν, ότι οποιαδήποτε επένδυση σε νέου αγωγού φυσικού αερίου και τερματικά δεν θα, μειώσουμε, δεν θα μειώσει την ε, προσπάθεια μετάβαση προ τι ανανεώσιμε και δεν θα μα οδηγήσει σε άχρηστα ε, στοιχεία ε, ενεργητικού για θέματα ενέργειας. Αντί να υποστηρίξουμε τέτοια έργα, δεν θα έπρεπε να υποστηρίξετε α, καθαρά project ενέργειας, αποκεντρωμένα, τοπικά, που λόγω του μικρού μεγέθους τους προφανώς δεν έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον κατάλογο εκεί. Μπορείτε να μου πείτε αν η Κομισιόν σκοπεύει να εισάγει μηχανισμούς για να ομαδοποιήσει διάφορα μικρά έξυπνα ε, project πράσινης ενέργειας και να τα υποστηρίξει. Και τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό ερώτημα, πότε θα κάνετε από πλευρά υπηρεσιών σας μία πλήρη διαφανή αξιολόγηση, ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ο τρέχον κατάλογος και ο επόμενο κατάλογος ΕΚΕ θα γίνει με βάση μια μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται στο ε, τρέχον πολιτικό πλαίσιο και στην ε, ενεργειακή ανάγκη που έχουμε και στι υποσχέσεις της Ursula von der Leyen να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση την πρώτη ήπειρο κλιματικά ουδέτερη. Τι σημαίνει αυτό. Ε, θέλουμε μια πολιτική πραγματικά στραμμένη προς το μέλλον που να είναι ρεαλιστική, αλλά να δράσουμε τώρα. Τελευταία παρέμβαση για να απαντήσει μετά η Επίτροπος, ο κύριος Τομισόφσκι. Με μικρόφωνο κατά ανάγκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας χαιρετώ, Επίτροπε, και εγώ. Κατά την παρουσίασή σας, σας είπατε ότι το φυσικό αέριο θα είναι και στο μέλλον σημαντικό. Ενώ θα ψάχνουμε λύσεις με υδρογόνο και βιοαέριο. Αυτό που βλέπουμε στην Ευρώπη είναι να παίρνουν αποφάσεις άλλε γενικές διευθύνσει που να κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις από αυτέ που μας λέτε εσείς. Ακούσαμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και μια άλλη τράπεζα επίσης λέει το ίδιο και η ΦΙΣΜΑ επίσης επικρίνει, τη στιγμή που επικρίνει το αέριο, λέει άλλα πράγματα. Έχουμε μια άλλη πρόταση, επίσης, με βάση την οποία υποτίθεται ότι μειώνονται οι ευκαιρίες για παραγωγή φυσικού αερίου. Αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, δεν εγκυμονούνται κίνδυνοι. Είναι μια πολιτική που υποσκάπτει το φυσικό αέριο και με αυτόν τον τρόπο δεν θα υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Πάντως οι μεν λένε τα, τα α, οι άλλοι λένε τα β. Πρέπει να συνομιλήσουμε μεταξύ μας οι διάφορες γενικές διευθύνσεις, τα διάφορα υπουργεία για να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση. Γιατί αυτό που συζητείτε, ας πούμε, στη δική σας γενική διεύθυνση δεν υποστηρίζεται από άλλες γενικές διευθύνσει. Αυτά. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις για την Επίτροπο. Έχουμε 10 λεφτά που θα μας διαθέσουν οι ερμηνείς μας. Να απαντήσετε σύντομα και συγκεκριμένα. Φυσικά έχουμε φιλόδοξου στόχου, θα προσπαθήσουμε να τους υλοποιήσουμε. Ε, ούτως ώστε το 2050 να είμαστε η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο. Αλλά βεβαίως χρειαζόμαστε επενδύσει γι' αυτό, για νέα δίκτυα και νέες διασυνδέσει. Για την ηλεκτρική ενέργεια, διασυνδέσει. Και κυρίω πρέπει να πούμε ότι ο κατάλογο ΕΚΕ, τα έργα κοινού ενδιαφέροντο, όπως αυτά τα, αυτή η διασύνδεση μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας και Πορτογαλίας είναι ακριβώς τέτοια. Επίσης η, η σύνδεση μεταξύ Γαλλίας και Ιρλανδίας, η Κελτική Συμφωνία. Είναι όλα αυτά έργα για διασύνδεση ηλεκτρική, για την ηλεκτρική ενέργεια. Αυτά τα έργα του καταλόγου μας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε περισσότερη πράσινη ενέργεια, περισσότερες, περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν όμως στον κατάλογο και έργα για το φυσικό αέριο, που επιτρέπει ας πούμε στην Πολωνία να διαφοροποιήσει τις οδούς ανεφοδιασμού της ε, σε φυσικό αέριο. Παραδείγματο χάρη, μία νέα οδός Πολωνία, Δανία, Νορβηγία. Είναι σημαντικό όλες οι περιφέρειες να έχουν τα εργαλεία για να μειώσουν σταδιακά τους ρηπαντές από τα ορυκτά καύσιμα και να αυξήσουν τις, ενεργειακές πηγές, τις πράσινες ενεργειακές πηγές. Γιατί όπως σας, είπατε, σας είπαμε, μετά το 2050 θα πρέπει να μηδενίσουμε το διοξείδιο του άνθρακα. Τώρα, κάποια συγκεκριμένα έργα. Γιατί δεν τα χρηματοδοτούμε πια. Έργα που ανήκαν στον τέταρτο κατάλογο. Έχουν κάποια έργα που συνδέονται με, το, με την επικράτειά τους κάποια κράτη-μέλη. Εμείς έχουμε μια διαφανή διαδικασία, το είπα και πριν, όπου τα κράτη-μέλη προτείνουν κάποια έργα. Υπάρχουν εμπειρογνώμονε εμπειρογνώμονες σε επίπεδο περιφέρειας και μας δίνουν τη γνώμη τους και έτσι είμαστε σίγουροι ότι καλύπτουμε όλες τις περιφέρειες. Τώρα πώς θα βοηθήσουν αυτά τα έργα τους καταναλωτές μας. Ακούστε και μια ανησυχία γι' αυτό. Πώς θα αντιμετωπίσουμε και θα εξαλείψουμε την ενεργειακή φτώχεια των πολιτών. Υπάρχουν και σήμερα λύσεις. Οι ψηφιακές πλατφόρμες, ας πούμε, που σε ορισμένε περιφέρειες βοηθούν τους καταναλωτές, τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να παρατηρούν σε ωριαία βάση την κατανάλωση ενέργειας και την τιμή που πληρώνουν. Και βοηθάει τους μικρούς παραγωγούς, που κάποια στιγμή είναι και καταναλωτές, να πουλήσουν την παραγωγή τους. Και η ψηφιοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο ε, για το μέλλον. Και στο μελλοντικό κατάλογο θα δούμε έργα με όλο και περισσότερο τέτοιο προσανατολισμό. Ακούστηκε μια ερώτηση γιατί μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο για τον τέταρτο ή τι θα συμβεί στον τέταρτο κατάλογο εκεί. Ελπίζω να τον εγκρίνεται αυτό τον τέταρτο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος. Με βάση την συνθήκη μπορεί να εκφράσει αντίρρηση για την θέση σε ισχύ τον, του καταλόγου αυτού με πλειοψηφία. Εάν συμβεί αυτό, τότε ο τρίτος κατάλογος, ο οποίος έχει 40% περισσότερα έργα φυσικού αερίου, θα παραμείνει ενισχύει περισσότερο από τον τέταρτο δηλαδή. Αυτό θα έχει αρνητικέ συνέπειε. Γιατί στον τέταρτο κατάλογο έχουμε πολλά νέα φιλικά προς το κλίμα έργα. Τρία, ας πούμε, έξυπνα δίχτυα ηλεκτρικής ενέργειας ή τέσσερα δίχτυα στη Σκανδιναβία Εάν δεν εγκριθεί ο κατάλογο, δεν υπάρχει επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση όμω αυτών των έργων. Ελπίζω να εγκρίνετε αυτόν τον κατάλογο. Και εγώ σα προσφέρω στενή συνεργασία από πλευρά μου κατά τη διάρκεια τη διαδικασία δημιουργία του πέμπτου καταλόγου. Thank you so much. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε και όλου του συναδέλφου που πήραν το λόγο. Έχουμε λοιπόν τη λίστα, όπως ε, μα εξηγήθηκε, μας εξηγήσατε. Ε, σε ό,τι αφορά την προσέγγιση αυτή η το ΜΑΠ έχουμε φυσικά και την ε, ε, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των συναδέλφων. Είναι απαραίτητο φυσικά ο κανονισμός αυτός να συνάδει με τους φιλοδοξούς στόχους μας. Και είμαι βέβαιος ότι αυτά δεν θα συνάδουν απαραίτητα με αυτά που θα παρουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Έιλερ είπε ότι θα πρέπει να έχουμε και μια ισορροπημένη προσέγγιση. Να έχουμε υπόψη λοιπόν πώς έχει σήμερα η κατάσταση και πώς αυτή η μετάβαση μπορεί να επιτευχθεί επιτυχώς. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, κυρία Επίτροπε. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Τα λέμε στην επόμενη συνεδρίαση. 22-23 Ιανουαρίου κατά πάσα πιθανότητα του 2020 του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. In January? <laughs>